of I think we should get started as our distinguished... Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Η αξιότιμη προσκεκλημένη μας, η Επίτροπος Τάισεν, έχει φτάσει. Ήρθε μετά από μια μεγάλη πτήση από την Ιαπωνία, κατευθείαν από το αεροδρόμιο. Φαίνεται όμως ολόφρεσκη. Να είμαστε λίγο έτσι καλοί μαζί της στις ερωτήσεις μας. Κυρία Επίτροπε, καλώς ήλθατε και να σας ε, καλωσορίσω θερμά στη σημερινή συνεδρίαση της, Επιστρο... της Επιτροπής Απασχόλησης. Νομίζω ότι όλα τα μέλη μας ε, ε, αδειμονούν αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουν μαζί σας σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο συντονισμός δεν είναι μόνο πολιτικά ευαίσθητος, όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά έχει και μεγάλη επίπτωση στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των θεσμών μας. Πρέπει να βρούμε λύσεις που θα επιτρέψουν στα θεσμικά μας όργανα να εγκρίνουν κανόνες με έναν ε, εύκολο και συντονισμένο τρόπο. Δυστυχώς οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να συμβιβαστούν για κάποια θέματα που παραμένουν ανεπίλητα και διχάζουν τα κράτη-μέλη όπως η εφαρμοστέα ε, νομοθεσία και η κύρωση. Θα υπάρξει μια παρουσίασή σας μετά ανταλλαγή απόψεων. Μετά ε, ελπίζουμε ότι θα διευκολυνθεί η λήψη απόφασης ε, για το αν θα συνεχίσει ή θα σταματήσει ε, η προσπάθεια να επιληθούν αυτά τα ανεπίλητα ζητήματα. Οι συντονιστές στην τελευταία του συνάντηση που έγινε στις 24 Ιουλίου 2019 συζήτησαν τις τρεις διαφορετικές επιλογές. Υπήρχε επιλογή 1 να γίνει επανέναρξη ολόκληρη της διαδικασίας από το 0. Η δεύτερη επιλογή είναι η ψηφοφορία στην Ολομέλεια είναι ήταν στις 19 Απριλίου του 19 και αναβλήθηκε. Ζητήθηκε ε, στις 20 Νοεμβρίου του 2008, βάσει της έκθεσης που τότε εγκρίθηκε από την Επιτροπή, να γίνουν κάποιες τροπολογίες και μετά να προχωρήσουμε σε μία ε, πρώιμη πρώτης ανάγνωση συμφωνία και η τρίτη επιλογή είναι να συνεχίσουν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις στο σημείο ακριβώς από το οποίο ε, από το σημείο ακριβώς στο οποίο σταμάτησαν και να συνεχίσουμε το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας του Μαρτίου του 2019. Εγώ πρότεινα η απόφαση των συντονιστών για το ποια επιλογή θα επιλέξουμε να ληφθεί μετά από τη συνάντησή μας μαζί σας. Έτσι λοιπόν οι συντονιστές θα συναντηθούν μετά από αυτό το θέμα για να συνεχίσουν τη συζήτησή τους σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό που σας έχουμε σήμερα εδώ και πραγματικά δημονούμε για τη συζήτηση. Οπότε, κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά μου να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα, να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Η Πρόεδρος ε, εξήγησε γιατί άργησα ελαφρώς. Όμως, να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ή την επανεκλογή σας πριν ξεκινήσω. Είναι χαρά μου που σας βλέπω εδώ και χαίρομαι που θα έχουμε και λίγες εβδομάδες μαζί να συνεργαστούμε πριν έρθει η νέα Επιτροπή. Η νέα κοινοβουλευτική θητεία είναι πάντοτε ένας, ε, είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος. Ε, με καλέσατε να έρθω να σας μιλήσω και το κάνω με χαρά. Στην τελευταία θητεία, Κοινοβούλιο, Κομισιόν και Συμβούλια έκαναν πολλές προόδους, εξυγχρόνισαν τους κανόνες. Ε, το εγχείρημα αυτό τελείωσε σχεδόν. Σχεδόν, όχι ακόμα. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ευκαιρία να πάρουμε μερικά από τα πιο σημαντικά κομμάτια των ανεπίλητων ε, ζητημάτων και να τα κάνουμε τα πρώτα επιτεύγματα του νέου κοινοβουλίου. Φαίνεται ότι το θέμα του συντονισμού στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης είναι πάρα πολύ τεχνικό. Ε, ε, θα ήταν όμως σημαντικό να επιληθεί γιατί θα άλλαζε η καθημερινή ζωή των πολιτών. Αυτό ισχύει στη δική μας περίπτωση γιατί ο συντονισμός αυτός θα κάνει την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων πραγματικότητα. Το δικαίωμα να ζει κανείς, να εργαστεί, να συνταξιοδοτηθεί οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα πιο πολύτιμα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Λίγοι όμως ασκούν αυτά τα δικαιώματα ε, και πρέπει πολλοί επίσης να αφήσουν ε, πίσω τους ε, δικαιώματα. Όταν ε, λοιπόν ένας πολίτης πηγαίνει από τη μία χώρα στην άλλη θα πρέπει να χάνει αυτά τα δικαιώματά του γιατί αυτά είναι το λιπαντικό στα γρανάζια της ελεύθερης κίνησης των προσώπων. Έτσι λοιπόν να πω ότι δεν θα εναρμονίσουμε, αλλά θα συντονίσουμε, θα διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες καλύπτονται από την νομοθεσία μιας χώρας κάθε φορά και θα πληρώνουν φορές σε αυτή τη χώρα μόνο. Επίσης, οι πολίτες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους ε, πολίτες της χώρας από την οποία καλύπτονται. Αυτό είναι βάση ε, της αρχής της μη διάκρισης που διέπει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από την αρχή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης η ΕΟΚ πριν από 21, 61 χρόνια ήδη είχε εγκρίνει κάποια τέτοια νομοθεσία και σήμερα πάνω από 70, από 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν σε μια χώρα διαφορετική από αυτή ε, που γεννήθηκαν. Αυτό συν ε, το 1,4 εκατομμύρια διασυνοριακούς εργαζόμενους και τους 8 εκατομμύρια αποσπασμένους εργαζόμενους αποτελεί το μεγάλο σώμα των εργαζόμενων εν κινήσει. Το σύστημα λοιπόν ε, της κοινωνικής ασφάλισης ε, και ο συντονισμός των συστημάτων είναι σημαντικά. Όταν ξεκινήσαμε με την Επιτροπή Juncker, τονίσαμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την δικαιοσύνη της εσωτερικής αγοράς. Έγινε προτεραιότητά μας να διασφαλίσουμε την συνεχή υποστήριξη της ελεύθερης διακίνησης προσώπων. Να έχουμε δίκαιους, ξεκάθαρους κανόνες. Δεν θα μιλήσω για όλες τις πρωτοβουλίες που πήραμε, αλλά είχαμε και την αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, επίσης τη δημιουργία της αρχής για την εργασία. Και όλα αυτά τα θέματα που σας εξήγησε σήμερα το πρωί ο Γενικός Διευθυντής, όλα αυτά ε, λόγω της ε, καλής συνεργασίας ε, με την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθαν εις πέρας και η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας αυτή τη στιγμή δημιουργείται αλλά και αναθεωρήθηκε και η οδηγία για τους αποσπασμένους επίσης. Τα κράτη-μέλη υποστήριξαν με μεγάλη πλειοψηφία αυτά τα δύο νομοθετικά κείμενα και αυτό δείχνει ότι είναι πολύ εύκολο, είναι δυνατόν μάλλον, να δημιουργήσουμε γέφυρες αυτά τα, σε αυτό το πλαίσιο προτείναμε τον εξυγχρονισμό των κανόνων για την κοινωνική ασφάλιση, διότι οι κανόνες θεωρούμε χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις για να είναι πιο εύκολο για τους εργαζόμενους, τους αναζητούντες εργασία και τις επιχειρήσεις να βρουν δουλειά και απασχόληση ε, καλή την πίστη, για να μπορούν όλοι να συνεργαστούν επικοδομητικά και να μην υπάρχει απάτη. Το Δεκέμβριο του 2016 έγινε η νομοθετική πρόταση. Φέτος, το Μάρτιο, μετά από 8 τριμερείς ε, διαλόγους, ε, είχαμε μια ισορροπημένη συμφωνία, όμως ε, δεν είχαμε την ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο που χρειάστηκε για να εγκριθεί αυτή, γιατί έλειπαν λίγες ψήφοι. Υπήρχαν πολλές και δυτικές και ανατολικές χώρες που υποστήριξαν την ε, ε, συμφωνία όπως και πολλές χώρες του Βορρά και του Νότου. Υπήρχαν ε, όμως κάποιες διαφορές μεταξύ των χωρών που στέλνουν ή δέχονται εργαζόμενους. Ελπίζω ότι με καλή την πίστη θα λύσουμε αυτά τα ζητήματα, ζητήματα και είμαι πεπισμένη ότι αν μπορέσουμε να συνεχίσουμε με έναν έντονο ρυθμό, η τελική συμφωνία θα είναι στο χέρι μας. Όσο πιο γρήγορα ξανά ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, τόσο το καλύτερο γιατί ο στόχος μας παραμένει σταθερός. Θέλουμε ξεκάθαρους, δίκαιους και εφαρμόσιμους κανόνες. Αυτές είναι και οι αρχές που υποστηρίζουν και όλα αυτά που ήδη έχουμε πετύχει στις ε, διαπραγματεύσεις. Έχουμε κλείσει δύο από τα τέσσερα κεφάλαια αυτό για τις μακροχρόνιες ε, παροχές και αυτό για τις οικογενειακές παροχές. Υπάρχει το θέμα των εργασιακών παροχών και της εφαρμοστές νομοθεσίας που αφορά στους κανόνες και στη διαδικασία που θα διασφαλίσουν ότι οι κινούμενοι πολίτες θα εμπίπτουν στη νομοθεσία μίας χώρας πάντοτε που ακόμα εκκρεμούν. Αλλά ακόμα και για αυτά τα δύο κεφάλαια φτάσαμε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε τη δουλειά που έπρεπε να γίνει. Ξέρετε πολύ από εσά ότι δεν φοβάμαι να πω ότι αυτά που πρότεινε αρχικά η Επιτροπή δεν ήταν τόσο καλά όσο οι λύσεις που βρέθηκαν τελικά από τους συνομοθέτες. Ο στόχος μου δεν ήταν ποτέ να κερδίσω πόντους, αλλά να βρω λύσεις για πρακτικά προβλήματα που θα ε, λάβουν την πλειοψηφία στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Με όλη μου την καρδιά λοιπόν θα υποστηρίξω οποιαδήποτε λύση που είναι καλύτερη από αυτή που προτείναμε, που είναι ξεκάθαρη, δίκαιη και εφαρμόσιμη. Έτσι φτάσαμε και ως εδώ και με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα που εκκρεμούν. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί θα προσφέρουν μεγαλύτερη ευκρίνεια και νομική βεβαιότητα όσον αφορά στις εργασιακές παροχές. Θα έχουμε συγκεκριμένους κανόνες για τη συσσόρευση. Επίσης, οι κινούμενοι πολίτες θα έχουν ε, την δυνατότητα για επιδόματα ενεργείας μόνο αν πληρούν τις ίδιες ε, προϋποθέσεις και κανόνες με, τη χώρα, με τους άλλους πολίτες της χώρας από την οποία καλύπτονται. Αν ένας, ε, ας πούμε, εργαζόμενος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον 300 ημέρες ε, για να μπορέσει να λάβει ταμείο ενεργείας, τότε αυτός ο κανόνας θα εφαρμόζεται και στους υπόλοιπους πολίτες της ίδιας χώρας που θα μετακινούνται στο, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το θέμα είναι ε, για την για τη συνταξιοδότηση, δηλαδή για τη συσσόρευση των δικαιωμάτων. Ε, ας πούμε, ε, όταν κάποιος θέλει να πάρει σύνταξη και επικαλείται ε, κάποιες προηγούμενες περιόδους εργασίας σε άλλες χώρες και θέλει αυτές να συμπεριληφθούν και να συνυπολογιστούν στη σύνταξή του. Τα, για τα ταμεία ανεργίας, τα κράτη-μέλη διαφορετικά εφαρμόζουν την αρχή. Οι συνομοθέτες πρέπει να βρουν λοιπόν ξεκάθαρους κανόνες. Αυτή την ευκρίνεια που χρειάζεται για να μπορούν τα κράτη-μέλη να έχουν μια συνεπή εφαρμογή των κανόνων. Οι αναθεωρημένοι κανόνες ορίζουν ότι περίοδοι προηγούμενη εργασία σε άλλη χώρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις αρμόδιες χώρες μέλη μόνο αν έχουν διαρκέσει παραπάνω από ένα μήνα. Έτσι λοιπόν έχουμε σαφήνεια και νομική βεβαιότητα αλλά και μεγαλύτερη δικαιοσύνη για τους κοινόμενους πολίτες και για τα κράτη-μέλη και τους φορολογούμενους πολίτες τους. Για παράδειγμα, για τους διασυνοριακούς ε, εργαζόμενους, όταν ε, υπάρχει δυνατότητα ε, καταβολής ε, ταμείου ενεργείας, ε, θα πρέπει να λεφθεί υπόψη που κατοικεί ο μεθοριακός υπάλληλος γιατί ε, ε, καταλαβαίνετε πως ε, το ένα κράτος θα έχει ευθύνε και όχι έσοδα και το άλλο ε, θα έχει έσοδα χωρίς ευθύνε. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν θέλει να το αλλάξει αυτό και να ε, συνδέσει τα δύο, δηλαδή τις ευθύνε με τα έσοδα. Πρέπει λοιπόν να πω ότι το Κοινοβούλιο έχει συμφωνήσει στο στόχο και στην αρχή ακόμα δεν έχουμε βρει τη λύση. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεθεί η λύση και θα είναι αποδεκτή και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο ως προς την Επιτροπή. Για άλλη μια φορά θα υποστηρίξει και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση είναι ξεκάθαρη, δίκαιη και εφαρμόσιμη. Τέλος, οι αναθεωρισμένοι κανονισμοί θα διευκολύνουν την καλύτερη εφαρμογή. Το θέμα της εφαρμογής είναι σημαντικό γιατί έχει να κάνει και με την ε, συνεπή ε, εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Αν θέλουμε να έχουμε ε, συνεχώς υποστηρίξη για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις καταχρήσεις και να διατηρούμε τις επιχειρησιακές ευκαιρίες των ε, εταιριών. Να ε, προστατεύουμε αυτούς που κινούνται, μετακινούνται, καλή την πίστη. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι αλλαγές που πρέπει έτσι ώστε ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης να εφαρμοστεί σωστά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εθνικά συστήματα να έχουν καλύτερα εργαλεία που θα μπορούν να τους βοηθήσουν να εξακριβώσουν τα στοιχεία. Αν ένας εργαζόμενος έχει εργαστεί σε πολλές χώρες ταυτόχρονα, μπορεί να χρησιμοποιεί το Α1, το φορητό έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την καταβολή εισφορών σε άλλο κράτος μέλος. Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί θα περιέχουν μια ξεκάθαρη διαδικασία. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες ε, για την ε, ε, διασφάλιση της ακρίβειας του εγγράφου και τον έλεγχο της ακρίβειας του εγγράφου και για να αποσύρονται τα πλαστά έγγραφα και με αναδρομική ισχύ. Επίσης, θα ξεκαθαρίζουμε οι κανόνες ότι δεν χρειάζεστε αυτό το έγγραφο για επιχειρηματικά ταξίδια και πολύ μικρές ε, μεταθέσεις, πολύ μικρής διάρκειας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το ε, έγγραφο για οποιαδήποτε, για οποιασδήποτε διάρκειας μετακινήσεις γιατί θα ήταν μεγάλη γραφειοκρατία και γενικά θα εμπόδιζε την άσκηση της ελεύθερης διακίνησης ε, εργαζομένων. Αυτά πρέπει να αναθεωρηθούν. Επί της αρχής αυτής έχουν ε, φυσικά συμφωνήσει ε, τα θεσμικά όργανα, απλώς δεν έχουν μπει οι λεπτομέρειες στο χαρτί θα πρέπει να το οργανώσουμε και η λύση είναι σχεδόν εκεί. Δεν έχω Δεν υπήρχε όμως αρκετός χρόνος να το εξηγήσουμε στα διάφορα κράτη-μέλη και υπήρξε μια μικρή ανασφάλεια από την πλευρά τους. Γι' αυτό δεν το δέχτηκαν ακόμα και πρέπει να το αποφασίσουν σε επίπεδο κορεπέρ. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο ορισμό του business trip, του επαγγελματικού δηλαδή ταξιδιού και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τη δράση που μπορεί να ληφθεί κατά των εταιριών, των επιχειρήσεων εκείνων που προσπαθούν να παρακάψουν του κανόνε. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που εργάζονται σε πάνω από μία χώρα και υπάρχουν και ορισμένε επιχειρήσει Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσει σε αυτό που προσπαθούν να αποφεληθούν τη κατάσταση αυτή. Δημιουργούν δηλαδή εικονικά, αν θέλετε, γραφεία προκειμένου να αναγκάσουν έναν εργαζόμενό του να υπαχθεί στο εθνικό εργατικό δίκαιο μια άλλη χώρα, ενώ στην πράξη δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Με τον αθεωρημένο κανονισμό θα έχουμε νέα κριτήρια προκειμένου να μπορούμε να παρακάμψουμε τα ψευδή αυτά πλαστά γραφεία και να μπορούμε πραγματικά να εχνηλατήσουμε την πραγματική πορεία του εργαζομένου και τους πραγματικούς χώρους εργασίας του. Και είμαι πεπισμένη ότι και στο ζήτημα αυτό θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Στη τελευταία ανάλυση είναι κοινό το συμφέρον μας να επιλύσουμε τα αυτά προβληματικά ζητήματα και θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες οι οποίοι να μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη προκειμένου να αποφεύγουμε αυτές τις απόπειρες παράκαμψης της ενωσιακής νομοθεσίας. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία εισηγήτρια, πριν από 60 χρόνια δημιουργήθηκαν οι κανόνες αυτοί ως βασικός κανόνας για να προωθηθεί η ελεύθερη κινητικότητα και η ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τους κανόνες αυτούς για τους εκατομμύρια πολίτες που ασκούν το δικαίωμα της κινητικότητας και σχεδόν έχουμε φτάσει στο επίπεδο αυτό. Αν συγκρίνουμε την κατάσταση με ένα ποδηλωτικό αγώνα, θα λέγαμε ότι περνάμε πλέον στην τελευταία φάση του αγώνα αυτού. Είναι πολύ σημαντικό όμω για να γίνει αυτό, για να ολοκληρώσουμε δηλαδή τον αγώνα, να ξεκινήσουν ευθύ αμέσω οι τριμερεί διάλογο μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση με την οποία θα συμφωνούμε όλοι. Θα ήθελα λοιπόν να σα στείλω το μήνυμα αυτό το οποίο προσπάθησα να διαβιβάσω και προ το Συμβούλιο και προ τα κράτη-μέλη δηλαδή. Δείτε πόσο πολύ έχουμε προχωρήσει, δείτε που έχουμε φτάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιδείξουμε τώρα την τελική αυτή βούληση για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να πετύχουμε το τελικό ευκταίο αποτελεσμά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη θέση για τυχόν ερωτήσεις. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. το που Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ εύκολο να δει κανείς πραγματικά πόσο προσιλωμένοι είστε προσωπικά στο ζήτημα αυτό και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όταν λέτε ότι ε, υπάρχουν ε, αρκετοί νέοι βουλευτές πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι έχουν αρχίσει να ανησυχούν ε, για την τροποποίηση του κανονισμού 883 του 2004, ένας κανονισμός ο οποίος είναι ιδιαίτερα τεχνικός, ο οποίος όμως έχει να κάνει πραγματικά με, την, με τους βαθύτερους στόχους, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κινητικότητα και την κυκλοφορία. Πρόκειται, αν δεν κάνω λάθος, για τον τρίτο ή τέταρτο κατά σειρά κανονισμό που έχει εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ζητήματα αυτά και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ πέρα ότι ο κανονισμός αυτός υπάγεται στο σύνολο ευρύτερων κοινοτικών κανονισμών που ακολουθούν την ίδια συλλογιστική και που έχουν ως στόχο να σημειωθεί πρόοδος σε ιδιαίτερα πολύπλοκα ζητήματα. Το σκέφτηκα καλά γιατί για μένα είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά Δύο χρόνια ολόκληρα εδώ στην Επιτροπή μας, Επιτροπή μας κάναμε τόση πολλή δουλειά ο εισηγητής και είναι σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, να δοθεί αξία σε αυτά που ήδη έγιναν και να μην αφήσουμε στην άκρη αυτό το τελευταίο βήμα. Και να πω ότι βάσει του ε, του παραδείγματος της ποδήλασίας να έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της διαδρομής. Ε, μας μένει ένα μικρό κομματάκι, αλλά αυτό είναι ανηφόρα. Πρέπει λίγο να ελέγξουμε τον εξοπλισμό μας ε, για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να ανέβουμε αυτή την ανηφόρα. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε λίγη προσπάθεια παραπάνω γιατί όλοι ξέρουν ότι αν δεν ανέβουμε αυτή την ανηφόρα θα χάσουμε την όθηση που κερδίσαμε ε, από τα προηγούμενα βήματα και δεν είναι και κανείς ευχαριστημένος με το status quo από ποια πλευρά και αν βρίσκεται. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε μια πολύ καλή προετοιμασία για αυτό το τελευταίο κομμάτι της δοκιμασίας. Έχουμε ήδη αναφέρει τα σημεία τριβής. Ξέρουμε όμως και πόσο σημαντική είναι η επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στους πόρους τους. Και αυτές οι τέσσερις ομιλίες ε, που θα μιλούσουν για την κοινωνική Ευρώπη, την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, ε, ε, σε αυτές τις τέσσερις κυριακάτικες ομιλίες θα πρέπει να βρούμε πραγματικά τα σημεία που θα μας βοηθήσουν να μην τιμωρήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην υποφέρουν από τα μειονεκτήματα αυτής της διαδικασίας. Είπατε ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση. Και θα κλείσω λέγοντας ότι το Κοινοβούλιο όταν κοιτάζει την ιστορία τα τελευταία χρόνια βλέπει ακριβώς ε, αυτό το ρόλο που έπαιξε ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων των κινούμενων εργαζομένων. Πάντοτε και σε συνεργασία με το Συμβούλιο προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και στο τέλος πάντοτε τα καταφέρνουμε. Μια λύση που θα ικανοποιεί όλους. Χαίρομαι λοιπόν για τη συνεργασία μας και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πολύ καλή προετοιμασία που έγινε για αυτό το τελευταίο κομμάτι της διαδικασίας. Ευχαριστήσουμε πολύ την εισηγήτρια η οποία πήρε πρώτη το λόγο, αλλά θα ακούσουμε συνεχεία τους συντονιστές και τους κοιόδης εισηγητές. Ο κανόνας εδώ πέρα είναι δύο λεπτά αγόρευση για τον καθένα σας, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλους συναδέλφους να πάρουν το λόγο, πέρα από τους τονιστές δηλαδή και τους πιο δυσηγητές. Ξεκινάμε με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Λέναρτς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρώτος. Σας δω συγγνώμη, σας δω συγγνώμη λέει πρόεδρος, είπα κυρία Λέναρτς. Κάνω συχνά το λάθος αυτό, σας δω συγγνώμη. Ο κύριος Λέναρτ λοιπόν έχει το λόγο και εξ ονόματος της ομάδας Renew Europe, ο κύριος Πισλάρου, αυτό το είπα σωστά. Είστε όντω κύριο. <laughs> Πολύ ωραία. Ετοιμαστείτε γιατί θα πάρετε το λόγο μετά τον συναδελφό σα από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Προσπαθώ με κάθε δυνατό τρόπο να συμβάλλω στην ισότητα των δύο φίλων, αλλά όχι με τέτοιο δραματικό αν θέλετε τρόπο. Να ευχαριστήσω την Επίτροπο Τάισεν για την παρουσία, παρουσία εδώ σήμερα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την μεταφορά που χρησιμοποίησε για τον ποδηλατικό αγώνα. Ξέρετε, στον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας όλα τελειώνουν με ένα ποτήρι σαμπάνια και όλοι ανακουφισμένοι που ο ποδηλατικός γύρος τελείωσε. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε εμείς να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Ξέρετε πολύ συχνά στα πλαίσια ενός αγώνα υπάρχει ένα συναγωνισμός και ανταγωνισμός. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς εμείς θα καταφέρουμε να φτάσουμε στην τελική γραμμή, στη γραμμή του τερματισμού όλοι μαζί ταυτόχρονα και όχι ένα μόνος του ξεχωρίζεται από τους άλλους. Σίγουρα τρία ολόκληρα χρόνια επεξεργαζόμαστε τον νομοθετικό αυτό φάκελο. Δεν είναι καινούργος λοιπόν. Ευχαριστήσουμε και τον πρώην εισηγητή μα, τον κύριο Γκυγιό Μπαλάσα, όλους τους συνεισηγητέ, συντονιστές, τις υπηρεσίες τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Κοινοβουλίου που κάνανε πραγματικά μια εξαιρετική εργασία όσον αφορά το φάκελο αυτό. Σαφώ η πρόταση αυτή δεν είναι καινούργια, αλλά έχει ανανεωθεί στο ενδιάμεσο διάστημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένω, κύριε Επίτροπε, Χρειαζόμαστε κι εμεί λίγο χρόνο προκειμένου να δούμε πώ διαμορφώνονται συζητήσει μεταξύ των πολιτικών ομάδων στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου, αλλά και με το Συμβούλιο τι επόμενε εβδομάδε και του επόμενου μήνε. Πάντω, συμφωνώ μαζί σα ότι ένα σημαντικό τμήμα τη εργασία έχει ήδη επιτευχθεί. Εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να εφεύρουμε εκ νέου τον τροχό σε όλα τα κεφάλαια. Ό,τι έχει συμφωνηθεί έχει ήδη συμφωνηθεί, μα ικανοποιεί. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τα ήδη συμφωνημένα κεφάλαια. Ανταυτού θα πρέπει να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο για να πετύχουμε την ευκταία ισορροπία για τα ζητήματα εκείνα τα οποία είναι προβληματικά και ακόμα εκκρεμούν. Και όπω είπαν και οι προαλήσαντε, οι κανόνε αυτοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί, επηρεάζουν εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Ο ίδιο προέρχομαι από μια παραμεθόριο περιοχή Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες ε, που και στη δική μου την εκλογική περιφέρεια παραπονιούνται για τους υφιστάμενους κανόνες. Νομίζω ότι κάλυψα τα δύο λεπτά που είχα στη διάθεσή μου. Ήθελα απλώς να σας πω ότι προσβλέπω σε μια πολύ θετική συνεργασία και με την εισηγητριά μας, την κυρία Μπίσοφ, και με τους σκιώδεις εισηγητές, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Άφησα περισσότερο χρόνο και τη αποκάλυψα κυρία. Η κυρία Λάγκετσίπε να προετοιμάζεται και τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπος του Renew Europe. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα πραγματικά και εγώ να σας συγχαρώ. Συμφωνώ και εγώ ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία από την αρχή. Θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας και αποφελούμε τις ευκαιρίες για να πω για μία ακόμη φορά ότι ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες μας εκλέγουν εδώ και σαφώς εμείς θα πρέπει να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντά τους για την ε, πολιτική ομάδα Renew Europe δεν θα μπορούσαμε να είχαμε πραγματική κινητικότητα ακόμα και ανταγωνιστική αγορά αν δεν υπάρχει συνεργασία και συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει να δίνουμε στους εργαζόμενους μας ε, τα δικαιώματα τα οποία έχουν στη χώρα τους και σε άλλες χώρες, στις οποίες ενδεχομένως να δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περίπου 5 εκατομμύρια Ρουμάνοι πολίτες ζουν εκτός Ρουμανίας και εργάζονται στις χώρες τις οποίες κατοικούν. Συμβάλλουν στην οικονομία των χωρών αυτών και εμπλουτίζουν, αν θέλετε, τι χώρε αυτέ και τι οικονομίε του με τι δεξιότητέ του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλου αυτού του πολίτε να καταφέρουμε να εγκρίνουμε το στομότερο δυνατό την νομοθεσία αυτή. Θα ήθελα να φωτίσω τρει πτυχέ. Πρώτον, υπάρχουν πολλοί εκ των πολιτών μα που προσπαθούν να κατοχυρώσουν τις παροχές τους αυτές για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή. Περνάνε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρουν πραγματικά να αποφεληθούν των παροχών αυτών. Το πρώτο μου λοιπόν ερώτημα είναι το ακόλουθο. Πώς μπορούμε μέσα σε 30 μέρες το ανώτερο να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα αυτά χωρίς να είναι απαραίτητο να ταξιδεύει κανείς κάποιος ενδιαφερόμενος στην χώρα κατοικίας του ή στη χώρα εργασίας. Δεύτερον, μακροπρόθεσμη φροντίδα, μακροπρόθεσμη θεραπεία. Πώς μπορούμε, μακροχρόνια περίθαλψη μάλλον, πώς μπορούμε να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στο δικαίωμα αυτό. Και τρίτον, πώς μπορούμε να εντοπίσουμε καλύτερες μεθόδους προκειμένου να γίνεται κάθε φορά η απαραίτητη τιμαριθμική αναπροσαρμογή και προκειμένου οι πολίτες πραγματικά να λαμβάνουν τα δικαιώματα και τις παροχές τα οποία δικαιούνται. Τώρα κυρία Λάγκεντζιμπεν και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Ζαμέ. Αγαπητοί επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζουμε φυσικά ε, το ότι πρέπει γρήγορα να κλείσει αυτό το θέμα. Υπάρχουν λίγα ακόμα εκατοστά που πρέπει να διανυθούν για να φτάσουμε ε, στο σημείο που πρέπει. Θα ήταν χαμένη ευκαιρία να μην κλείσει το θέμα τώρα. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι και είναι και για μας ε, σημαντικό αλλά και για την Επίτροπο και φυσικά για τους πολίτες. Μετά από τρία χρόνια εργασίας σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, θα ήταν καταστροφή. Επίσης, ε, ε, να ξέρετε ότι δύο με τρία χρόνια χρειάζονται για να εφαρμοστεί μια διαδικασία και πραγματικά αυτό μπορεί να μην φαντάζει πολύ, αλλά φαντάζει τεράστιο διάστημα για έναν πολίτη ο οποίος ε, χρειάζεται να ταξιδέψει ή να εργαστεί στο εξωτερικό. Θα πρέπει λοιπόν ο συντονισμός αυτός να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται και είναι πολύ σημαντικό. Ας είμαστε πραγματιστές. Ξέρω ότι αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες ε, δυνάμεις μας, όπως είπε και η Επίτροπος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ε, να εργαζόμαστε σκληρά για να μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία ε, και πραγματικά όταν η ε, γερμανική κυβέρνηση στο Συμβούλιο σταματήσει να βάζει φρένο σε όλα αυτά, θα θυμηθούν οι πολίτες ποια είναι η Ενωμένη Ευρώπη ε, αλλά δυστυχώς επειδή τα πράγματα έχουν ε, γίνει έτσι ως τώρα δεν μπορώ να το εγγύθω. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την κυρία Ζαμέ και μετά η κυρία Ρατοκόσκα. Κυρία Ζαμέ. Δεν είναι εδώ η κυρία Ζαμέ. Η κυρία Ραφάλσκα. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να πω ότι μας ικανοποιούν τα κεφάλαια που αφορούν την ίση μεταχείριση και τα οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ενεργείας και άλλες παροχές. Είπατε κυρία Επίτροπη ότι οι λύσεις που προσφέρονται εδώ είναι καλύτερες από αυτές οι οποίες είχαν προταθεί αρχικά. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και πολλές αμφιβολίες και ενδιασμοί όσον αφορά κάποια βασικά θέματα. Αυτό κυρίως αφορά τους ε, αποσπασμένους ε, εργαζόμενους σε κάποια άλλη χώρα. Έχω μία ερώτηση που αφορά τα νέα κριτήρια για τις χρονικές περιόδους και που αφορούν τον τζίρο των επιχειρήσεων ή τον κύκλο εργασιών τους ή τα κέρδη τους, που είναι παράγοντες οι οποίοι πολλές φορές καθορίζουν περισσότερο από τους κανόνες για όρους στην νομοθεσία. Αυτό αφορά ίσως κάποιους ε, εργαζόμενους σε ειδικού τομείς, τον οικοδομικό ή άτομα τα οποία φροντίζουν κάποια άτομα ασθενή. Εδώ έχουμε πολλές αμφιβολίες και έχουμε και έναν ανοιχτό κατάλογο κριτηρίων, άρα μπορούν να προσθεθούν και άλλα κριτήρια. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Αναφέρατε το έντυπο αναφέρεται και το θέμα της απάτης και βεβαίως με πρόσθετη γραφειοκρατία ξέρουμε ότι δεν λύνονται πάντα τα προβλήματα της απάτης. Ο κύριος Μποτέγκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις που κάνατε, για την, για την παρουσίασή σας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην Ευρώπη. Ότι είναι καλό να μην το ξεχάσουμε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι συνάντησα κάποιον ο οποίος εργάζεται στον τομέα των οπροκυπευτικών και μου είπε ότι εγώ ζω και δουλεύω σε πολύ πρόσκαιρες συνθήκες, επισφαλής. Κάτι θα πρέπει λοιπόν να γίνει. Με ρώτησε, μπορεί να κάνει για μένα κάτι η Ευρώπη. Εσείς που είστε στην, ε, Βρυξέλλες μπορείτε να κάνετε κάτι. Βεβαίως, είπα εγώ. Μπορούμε να ασχοληθούμε με το θέμα των κοινωνικών παροχών και να εξασφαλίσουμε το ότι από την πρώτη μέρα της εργασίας του ο κάθε εργαζόμενος θα συμμετέχει στα κοινωνικά συστήματα ώστε να έχει και κοινωνικές παροχές. Το κείμενο λοιπόν στη θεωρία μπορεί να προσφέρει τέτοιου είδους δυνατότητες αλλά τώρα έχουμε χαθεί κάπως στις διάφορες συζητήσεις με τις χρονικές περιόδους. Γιατί να μην προβλέπετε κάτι από την πρώτη μέρα που εργάζεται κάποιος. Στην παρουσίασή σας επίσης, πολλές φορές αναφερθήκατε στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να παρεμποδίσουμε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή την ελεύθερη διακίνηση. Δεν θα πρέπει όμως να δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα στα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε, γιατί διαφορετικά τι μπορείτε να κάνετε. Τελειώσαμε με τον πρώτο γύρο ερωτήσεων της εισηγήτριας και των σχεδόν εισηγητών. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην Επίτροπο για να απαντήσει και μετά θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων για όλα τα άλλα τα μέλη που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ε, ένα λεπτό ο καθένας στη διάθεσή του, γιατί είστε πάρα πολλοί αυτοί που θέλετε να λάβετε το λόγο. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε σας. Ευχαριστώ όλους. Πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια και όλους τους σκιώδες εισηγητές που έλαβαν το λόγο. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα διότι υποστηρίζετε και αναγνωρίζετε την εργασία που έχουν κάνει οι συναδελφοί σας και στο παρελθόν για να γνωρίζετε το ότι έχουμε καλή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Είπατε, κυρία Σιγήτρια, ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα και μπορούμε να προχωρήσουμε βάσει αυτή τη δουλειά που έχει επιτελεστεί. Όπω είπε και στην Ολομέλεια σα σήμερα το πρωί ο Γενικό Διευθυντή, είμαστε στη διάθεσή σα, αν θέλετε περαιτέρω εξηγήσει τεχνική υποστήριξη για να καταλάβετε περί τίνο πρόκειται. Διότι όντω πρόκειται για κάτι το τεχνικό και πολλέ φορέ χρειάζεστε εξηγήσει ε, για να από μένα ή κάποιον ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα και μπορεί απλά να σας εξηγήσει. Να συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε με εξαιρετικό τρόπο όπως κάναμε μέχρι τώρα. Τώρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λέναρτς για τις παρατηρήσεις που έκανε. Ελπίζω ότι μπορούμε μεταξύ συντονιστών να συμφωνήσουμε για να ξαναρχίσουμε να δουλεύουμε. Γιατί πρόκειται μια δουλειά πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις και θα προσπαθήσω το συντομότερο δυνατό να τις απαντήσω. Πώς να εξασφαλίσουμε, όπως είπε ο κύριος Πισλάρη, κυρία Πισλάρη, συγγνώμη, ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ωφέλη για τον εργαζόμενο, αλλά γιατί από την 30η μέρα και μετά. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες και από νομικής πλευράς την βεβαιότητα ότι όλοι θα γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Είναι εδώ ο κύριος Λέναρτς και έκανε την ίδια ερώτηση. Τι θα μας βοηθήσει πολύ οι εθνικές αρχές των κρατών μελών να συνεργαστούν να συνεργάζονται καλύτερα από ό,τι έκαναν μέχρι τώρα, διότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, διότι θα δημιουργηθεί μία καλύτερη συνεργασία από την στιγμή την οποία όλοι τα, όλα τα υπεύθυνε αρχές όλων των κρατών μελών θα συνεργαστούν για να μπορέσουν να διασταυρώσουν πληροφορίες και να λύσουν καλύτερα τα προβλήματα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχει υποχρέωση να απαντούν οι αρχές σε επιστολές, να δίνουν εξηγήσει. Αλλά δεν υπάρχουν προθεσμίες και εδώ θα πρέπει να βάλουμε προθεσμίες. Προθεσμίες ε, αρκετά σε λίγες ημέρες, ώστε να μπορεί κανείς να περιμένει την απάντηση που περιμένει ε, αρκετά σύντομα, αλλά να είναι σαφείς και οι απαντήσεις οι οποίες του δίνονται για να καταλαβαίνει πώς θα προχωρήσει. Πίσω λοιπόν στα πλαίσια τριμερούς διαλόγου θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Όταν αφορά τα ο, νιατρική περίθαλψη τα ωφέλη για μακροχρόνιες τέτοιου είδους θεραπείες. Υπάρχει νομοθεσία και η νομολογία λέει ότι τέτοιου είδους προβλήματα θα πρέπει να επιλύονται όπως επιλύονται τα προβλήματα που αφορούν μία ασθένεια οποιοδήποτε. Και βεβαίως υπάρχει και νομοθεσία. Αλλά το ερώτημα είναι να ορίσουμε τι είναι ιατρική φροντίδα μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε σαφείς ορισμούς στη νέα νομοθεσία. Στα πλαίσια λοιπόν του τριμερούς διαλόγου έχουμε ορισμό και θα υπάρχει στο παράρτημα κατάλογος ο οποίος θα συμφωνηθεί λεπτομερώς μεταξύ κρατών μελών ώστε να μπορούν και οι πολίτες και οι εθνικές αρχές να ξέρουν ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα δικαιώματα των οποίων χαίρουν και σε άλλες χώρες. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο σύστημα και ένα ενιαίο έγγραφο ενδεχομένω. αν αυτό ε, μπορεί να είναι πιο λειτουργικό και καλύτερο, διότι έτσι θα μας βοηθήσει να λύσουμε πολλά προβλήματα. Χαίρομαι για την υποστήριξη εκ μέρους των ε, σκιώδους εισηγήτριας εκ μέρους των Πρασίνων στο Συμβούλιο συζητούμε και με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της Φινλανδικής Προεδρίας και νομίζω ότι θα επιτευχθεί και σε αυτό το επίπεδο πρόοδος. Στην κυρία Ραφάλσκα από την ECR θα πω ότι χαίρομαι διότι τα περισσότερα κεφάλαια είπατε ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση Βεβαίω θα πρέπει να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Το κάνουμε αυτό ώστε οι προτάσεις να είναι νομικά σωστές και να καλύπτουν τον τρόπο. Επίσης έχουμε το θέμα των απασχολούμενων συγχρόνως σε πολλά κράτη-μέλη. Και το ερώτημα είναι πού ανήκουν. ο συντονισμός των κοινωνικών συστημάτων είναι η ενότητα. Δηλαδή, σε μία χώρα είναι ενιαίο το σύστημα, αλλά πρέπει να, να δούμε για αυτούς τους εργαζόμενους ε, πού καταβάλει την κοινωνική του εισφορά εργαζόμενος και πού ε, απολαμβάνει των υπηρεσιών και των όφελων. Φαίνεται πολύ τεχνικό αυτό που σας λέω, δεν είναι όμως τόσο πολύ τεχνικό. Εάν ένας εργαζόμενος εργάζεται σε περισσότερο από ένα κράτος μέλος και έχει μία δραστηριότητα στον τόπο κατοικίας του, εάν δηλαδή εργάζεται περισσότερο από το 25% του χρόνου εργασία του, η χώρα αυτή είναι η χώρα η οποία έχει για την ε, κοινωνική ασφάλιση την αρμοδιότητα. Τώρα εξαρτάται και από πού ποια είναι και η έδρα της επιχείρησης για την οποία εργάζεται. Ποια είναι η πραγματική έδρα της επιχείρησης. Πολλές φορές είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε και εδώ κριτήρια που θα μας βοηθήσουν να θεσπίσουμε σαφείς κανόνες με πολύ ισχυρή νομική βάση και να ξέρουμε βάσει των κριτηρίων που δραστηριοποιείται περισσότερο η τάδε επιχείρηση κριτήρια τα οποία θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και όλοι να τα χρησιμοποιούν και να βασίζονται σε αυτά. Ακόμη είμαστε σε επίπεδο συζητήσεων και θα πρέπει πραγματικά να συντονιστούμε. Και να δούμε ποια στοιχεία χρειαζόμαστε ώστε να υπάρχει η νομική βεβαιότητα, να αποφύγουμε τις απάτες και να έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα. Ένα σύστημα που να λειτουργεί υπέρ των πολιτών, των επιχειρήσεων και ένα σύστημα το οποίο θα μπορούμε να ε, χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. Ένας άλλος συναδελφός σας μας μίλησε για τον εργαζόμενο ε, εποχιακά στον τομέα των λαχανικών. Ποια είναι η κυρία δραστηριότητα αυτού του εργαζόμενου πώς μπορεί να προστατεύεται πάλι ο εργαζόμενος. Και όπως είπα και στην κυρία Ραφάλ, εάν το 25% της επαγγελματική δραστηριότητας είναι πάνω από το 25% σε μια χώρα, αυτή η χώρα είναι υπεύθυνη για τα κοινωνικά θέματα και την κοινωνική προστασία του εργαζόμενου. Επίσης, αν εργάζεται σε μια επιχείρηση, όπως και προηγουμένως, πρέπει να δούμε πού είναι η πραγματική έδρα της επιχείρησης. Προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου ασχοληθήκαμε επίσης με θέματα κοινωνικής ασφάλειας. Και τώρα θα πρέπει να δούμε όταν έχουμε αποσπασμένους εργαζόμενους, ένα εργαζόμενο που μετακινείται για να εργαστεί σε μια άλλη χώρα και έχει μια σύμβαση με έναν εργοδότη εκεί, ο εργαζόμενος αυτός πρέπει να την χάνει της ίδιας μεταχείρισης που την χάνουν οι εργαζόμενοι της χώρας στην οποία πηγαίνει. Ο ίδιος εργασιακός κώδικας, η ίδια κοινωνική ασφάλεια, οι ίδιες παροχές, η ίδια συνεισφορά. Όταν κάποιος μιλάει όμως για αποσπασμένο εργάτη, ε, εργαζόμενο, συγγνώμη, έχουμε να κάνουμε με κάποιον ο οποίος προσωρινά πάει σε μια άλλη χώρα. Θα πρέπει όμως όπως έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες μας, για όλους αυτούς τους εργαζόμενους να εξασφαλίζουμε τις υποχρεώσεις και δικαιώματα. Όταν κάποιος είναι αποσπασμένος για μικρό χρονικό διάστημα, ίσως δεν μπορούμε να τα συγκεράσουμε όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τα κοινωνικά δικαιώματα και τις παροχές του αποσπασμένου. Ποια χρονική περίοδο? Κάποιους μήνες, ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο δύο χρόνια όταν υπάρχει αλλαγή της νομοθεσίας. Γι' αυτό χρειαστήκαμε τόσο καιρό ώστε να μπορέσουμε να συγκεράσουμε όλα αυτά τα θέματα και να, να καταλήξουμε σε συμφωνία ώστε να ξέρουν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι τι σύστημα ακριβώς θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων πολύ θέλετε να πάρετε το λόγο. Ο κύριος Κώσα και ας ετοιμάστε και ο κύριος Σμίτ. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα και ουσιαστικά σας παραχωρώ και περισσότερο χρόνο γιατί τοποθετήθηκε πολύ γρήγορα η Επίτροπος αφήνοντάς μας έτσι λίγο περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, τα τελευταία τρία χρόνια πολλές φορές συζητήσαμε αυτή την πρόταση, καταφέραμε να φτάσουμε σε συμφωνία. Η Ουγγρική αντιπροσωπεία του ΕΛΚ ε, δεν ζήτησε συγκεκριμένα συντονισμό όμως ε, ε, πραγματικά βάσει ε, των όσων έχουν γίνει, υποστηρίζουμε τον καλύτερο συντονισμό. Νομίζω λοιπόν ότι η νέα κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιμετωπιστεί με τρόπο που να μην δημιουργήσει προβλήματα. Είμαστε σε προβληματική κατάσταση και χρειαζόμαστε χρόνο στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν ώστε να σκεφτούμε ακριβώς πώς θα δράσουμε. Ε, όταν έρθει και η νέα επιτροπή, ο κύριος Σμιτ και η κυρία Σάντερ παρακαλώ να ετοιμαστούν. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, να υπογραμμίσω τη σημασία αυτού του κανονισμού και την πραγματική πρόοδο που έχει γίνει και που είναι σημαντική και για τους εργαζόμενους και για την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας. Το βασικό πρόβλημα που απομένει είναι το θέμα των μεθοριακών εργαζόμενων. Όντως, ε, το να βρούμε ε, λύσεις ε, που είναι ισότιμες ε, και για αυτούς ε, τους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους για να έχουν, ε, να έχουν και αυτοί λοιπόν ένα δικαίωμα να βρουν εργασία υπό σωστές συνθήκες εκεί που διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους. Τώρα, για τον καταμερισμό του κόστους. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, σας θυμίζω, μια λύση. Υπάρχει η επιστροφή των πέντε μηνών του Ταμείου Ενεργείας. Επίσης, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις ικανότητες του κάθε κράτους μελούς να διασφαλίζουν σε όσους χάνουν τη δουλειά τους και πρέπει να βρουν καινούργια τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες με το νέο σύστημα ε, αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να διατηρηθεί. Έτσι να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, τις καλύτερες υπηρεσίες ε, και να βοηθήσουμε έτσι ώστε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την απάτη και την κατάχρηση. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει περιθώριο να εμβαθύνουμε. Η κυρία Σάντερ και η κυρία Ραφαέλα παρακαλώ. Merci, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω εδώ. Εργαστήκαμε μαζί με δική σας πρωτοβουλία για πέντε χρόνια προκειμένου να προωθήσουμε περισσότερο την κοινωνική Ευρώπη. Για το συγκεκριμένο μου ζήτημα Δυστυχώ δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο ευκταίο αποτέλεσμα, δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τι συζητήσει και αυτό είναι πραγματικά κρίμα. Ωστόσο νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε εκ νέου πολύ γρήγορα τις εργασίες μα χωρί όμω να ξεκινάμε από το μηδέν. Α μην το ξεχνάμε, έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε αξιοθαύμαστη πρόοδο σε πάρα πολλά κεφάλαια και νομίζω ότι λίγο μας μένει ακόμα για να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το νομοθετικό αυτό φάκελο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στις παραμεθόρειες περιοχές και κυρίως στους μεθοριακούς εργαζόμενους, γιατί είναι ακριβώς στις περιοχές αυτές που δημιουργούμε την Ευρώπη, που βιώνουμε την Ευρώπη σε καθημερινή βάση. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο σαφώς να βοηθήσουμε τους μεθοριακούς εργαζόμενους, αλλά και τις ίδιες επιχειρήσεις οι οποίες διαστηνοριακά και μεθοριακά φροντίζουν να παρέχουν υπηρεσίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε λοιπόν την απαραίτητη λύση για να έχουμε δικαιώματα τα οποία θα είναι δίκαια και ισότιμα για όλους. Η κυρία Ραφέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, αλλά και για την προσήλωση που δείχνετε για το ζήτημα αυτό. Η Επιτροπή Γιούνκερ ήδη από τις απαρχές της είχε πει ξεκάθαρα ότι θέλει να ασχοληθεί με τα μεγαλεπίβολα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τόσο πολύ με τα προγράμματα ίσονος σημασία. Εδώ αναφερόμαστε όντως σε ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, απασχόληση, σταθερή απασχόληση και σταθερό εισόδημα. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο κατεπολεμούμε την ένδυα, μόνο κατά αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνουμε ισότιμες ευκαιρίες για όλους. Τα δικαιώματα λοιπόν αυτά, οι ευκαιρίε αυτέ θα πρέπει να κατοχυρώνονται και μέσω τη νομοθετική αυτή πρόταση. Από κοινού λοιπόν πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο. Προσεγγίζουμε τα ζητήματα από την ίδια οπτική γωνία, θεωρώ, και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Παρ' όλα αυτά όμω, ποιο μήνυμα θα διαβιβάσετε στον διάδοχό σα αυτόν που θα σα διαδεχθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι άνθρωποι στι κάτω χώρε απαιτούν μεγαλύτερη σαφήνεια αυτή τη στιγμή για το τι θα ισχύει στο μέλλον όσον αφορά τα συστήματα κοινωνική ασφάλισης. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε και από εσά μια δέσμευση προκειμένου να ζητήσουμε από τον διάδοχό σα να τηρήσει τη δέσμευση αυτή. Ο επόμενο ομιλητή, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την όλη εργασία που έχετε επιτελέσει, για τη σημαντικότατη αυτή πρόταση κανονισμού και για όλη την εργασία που έχει επιτευχθεί υπό την επίβλεψή σας από το 2016 μέχρι και την περασμένη Άνοιξη. Είμαι πεπισμένη ότι Όλα τα επιτεύγματα αυτά θα οδηγήσουν σε βελτίωση τη ζωή και του βιωτικού επίπεδου των Ευρωπαίων πολιτών. Και όπω είπαν και οι προλαλήσαντε, ο προτινόμενο αυτό κανονισμό σαφώ θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να ανταποκρίνεται πλέον στι νέε προκλήσει που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια, από τότε δηλαδή που είχαμε την τελευταία αναθεώρησή του μέχρι σήμερα. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία να καταφέρουμε να προωθούμε περισσότερο την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών και να πόκειται στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπούν άλλωστε του Ευρωπαίου πολίτε, από κοινού να καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον το οποίο να είναι δίκαιο και ισότιμο για όλου του Ευρωπαίου οι οποίοι εργάζονται εκτό τη χώρα του. Προκειμένου όμω να καταλήξουμε σε μια κοινή βάση, θα πρέπει να επιτευχθούν σημαντικοί συμβασμοί από όλε τι πλευρέ. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγούμε λίγο από τα χαρακόμματά μα, θα πρέπει ενδεχομένω να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μα. Ποια είναι η άποψή σα, κύριε Επίτροπο, όσον αφορά τη στάση του Συμβουλίου. Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία της του προτινόμενου αυτού κανονισμού που αν αρθούν θα οδηγήσουν το Συμβούλιο σε ένα συμβασμό. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να κινηθεί λίγο περισσότερο το Συμβούλιο. Η κυρία Φερνάνδη έχει το λόγο και σε ετοιμάζεται και ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για την παρουσία σας. Είμαστε εδώ, εδώ ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων και όποιος εργάζεται σε άλλη χώρα να το κάνει με αξιοπρεπή τρόπο και να προστατεύεται. Είναι δικαίωμα η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, είναι θεμελιώδες δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών. Όπως είπατε όμως, ήδη έχουν γίνει στη διάρκεια της θητείας προηγούμενης πάρα πολλές ε, ε, έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος, παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες γκρίζες ζώνες και έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται με επισφαλείς πρόσκαιρες συνθήκες και πολλές φορές ε, είναι ανενημέρωτοι ή αποτελούν αντικείμενο απάτης. Πολλές φορές τα δικαιώματά τους τα βασικά καταστρατηγούνται ή υφίστανται διακριτική μεταχείριση. Θα πρέπει λοιπόν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε αυτό τον σημαντικό πυλώνα της εσωτερικής αγοράς ίσης όρης για όλους να προχωρήσουμε. Όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο και την Επιτροπή ε, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μία πάρα πολύ εκτενή και δύσκολη διαπραγμάτευση. Οι σοσιαλιστές στην Ισπανία θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να υπάρχει μία σωστή ε, συμφωνία για αυτά τα θέματα για να μην λώσουμε, δώσουμε λάθος μηνύματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Κυρία Σατόρη, αγαπητοί Επίτροποι, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μας απασχολεί σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αλλά πολλέ φορέ αποτελεί διακείμενο πολιτική εκμετάλλευση από κάποιε χώρε. Όπω δυστυχώ και στη χώρα μου. Ευρωπαϊκό συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλισης είναι ευρωπαϊκή πρόκληση. Θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσει στο κείμενο σύστημα. Δεν είναι ίσως πάντα αυτό το τελειότερο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε τους προστατευτισμούς και να έχουμε ένα ισχυρό σύστημα προστασίας του εργασμένου για όλους. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε περιπτώσεις όπως αυτές της Φλαμονβίλ και την εκμετάλλευση Γάλλων και Ρουμάνων εργαζομένων σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ε, συμπολιτών μας και να μην επιτρέψουμε στους λαϊκιστές να προτείνουν ε, κάποιους κανόνες οι οποίοι δεν είναι κανόνες δίκαιοι. Δεν είναι ώρα να λέμε αυτοί εναντίον ημών, αλλά όλοι μαζί με πνεύμα ευρωπαϊκό να συντονιστούμε για να προχωρήσουμε. Εγώ Πάρω τώρα εγώ το λόγο και έπειτα ο κύριος Βίλμς. κύριε Επίτροπε, καθότι αυξάνεται όλο και, μεγα... όλο και περισσότερο αριθμό των πολιτών οι οποίοι κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάζονται στο εξωτερικό, εκτός της χώρας τους δηλαδή, πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις νέες αυτές ανάγκες ο νέος αυτός κανονισμός, πώς μπορούμε να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις χωρίς να δημιουργήσουμε ιδιαίτερα υψηλό διοικητικό άχθος. Θα πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένε εξαιρέσει, ιδίω όσον αφορά τις περιπτώσεις των επαγγελματικών ταξιδιών business trips. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιούμε ευρέω το έντυπο Α1 και τι θα γίνει με, την, με τον τόπο εκείνο που θα πρέπει οι εργαζόμενοι να καταβάλουν τις εισφορές τους στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος πάλι, σας ζητώ σε συγγνώμη. Κύριε να έχετε το λόγο και κυρία Φράνσεν, εν συνεχεία. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως όταν βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας. Ωστόσο, τα όσα προβλέπονται αυτή τη στιγμή για τις παροχές ενεργείας από την πρόταση αυτή κανονισμού ενδεχομένως να μην λειτουργούν υπέρ των πολιτών και μπορεί να έχουν και κάποιες δυσμενείς ακόμα επιπτώσεις. Όπως θα ξέρει και η Επίτροπος, Διαφέρουν πάρα πολύ από τη μία χώρα στην άλλη τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Οργανώνονται με διαφορετικό τρόπο. Σε ορισμένε χώρες έχουμε υψηλό επίπεδο παροχών ανεργίας, όπου απαιτείται όμως και υψηλή χρηματοδότηση των εν λόγω ταμείων. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα στη Δανία, τη δική μου τη χώρα, χώρα στην οποία μπορούν οι πολίτες οικειοθελώς να συνεισφέρουν στο Ταμείο Ανεργίας, με προσωπική δηλαδή συνεισφορά τους, προκειμένου να μπορούν εν συνεχεία να αποφεληθούν από τα Ταμεία Ανεργίας και στην περίπτωση αυτή μπορούν να έχουν ένα υψηλό επίπεδο παροχών ανεργίας για μια περίοδο δύο ετών. Αυτό διαφέρει πολύ θεωρώ από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το σύστημα ανεργίας σε άλλες χώρες και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε και πάρα πολλές αποκλήσεις από τη μία χώρα στην άλλη. Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση εκείνη που θα έχουμε εργαζομένους από άλλες χώρες, οι οποίοι εργάζονται στη Δανία και οι οποίοι όμως δεν θα συνεισφέρουν στο δικό μας το σύστημα και παρόλα αυτά όμως θα έχουν απαιτήσει παροχών από το δικό μας Ταμείο Ενεργείας. Δεν θεωρείτε ότι κατά αυτόν τον τρόπο βαθμία θα, αρχίσουμε να, θα αρχίσει να μειώνει το αριθμό των πολιτών εκείνων που συνεισφέρουν στα ταμεία ενεργείας και αυτό ουσιαστικά δεν θα θέσει να αμφιβόλο την ίδια τη βιωσιμότητα των ταμείων αυτών η κυρία Φράνσεν και ο κύριος Μπεργλές στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι σήμερα μιλάμε όντας το ίδιο μήκος κύματος οι περισσότεροι. Θα ήθελα λοιπόν να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική αξιέπαινη εργασία που έχετε κάνει για το ζήτημα αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι θα πρέπει η τελική συμφωνία να είναι καλά ισορροπημένη. Στο πλαίσιο λοιπόν της όλης διαδικασίας θα πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα όσον αφορά το ζήτημα του συνυπολογισμού των δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις υπερβολές. Ξέρετε το βελγικό πλαίσιο, γνωρίζετε ποιες είναι οι βελγικές ευαισθησίες. Θα πρέπει να συζητήσουμε και πολλές εναλλακτικέ μεθόδους όσον αφορά το ζήτημα της επιβολής του κανονισμού αυτού. Θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να ισχύουν και συγκεκριμένε προθεσμίες όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και ένα σύστημα κοινοποίηση το οποίο να είναι ευκόλως προσβάσιμο αλλά και ευχριστό. Μέχρι στιγμής παρακολουθούσα το ζήτημα αυτό σε εξωτερικός παρατηρητής. Αυτή τη στιγμή αρχίζω και ανήκω και εγώ στην ομάδα εργασίας και διαπραγμάτευσης και πραγματικά σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το εξαιρετικό έργο το οποίο έχετε κάνει. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είμαι νέος Ευρωβουλευτής και ειλικρινά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη σημαντικότητα εργασία που έχετε ήδη επιτελέσει και να σας στείλω και ένα μήνυμα θα ήθελα να διαβιβάσετε δυνατόν το μήνυμα αυτό στη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι πρέπει πάση θυσία να επιταχύνουμε την εργασία την οποία κάνουμε για την νομοθετική αυτή πρόταση. Θεωρώ ότι είναι εξέχουσα σημασίας όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της, αλλά και προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις εκκρεμείς προκλήσεις που υφίστανται για την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Ακόμα και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του αποκλεισμού ορισμένων Ευρωπαίων πολιτών από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ακόμα και για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του αποκλεισμού των μεταναστών που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ισχύουν ισότιμοι κανόνε για όλου. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να υπερασπίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σταθούμε κατά οποιασδήποτε απόπειρα γίνεται για να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες, ιδίως και για την χρησιμοποίηση των κοινών αυτών μεθόδων και εντύπων που αναφερθήκατε. Κυρία Γκέμα, σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρέπει να θυμηθούμε ότι το ζήτημα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και του συντονισμού τους και το λέω αυτό από προσωπική πείρα, είναι ένα ζήτημα το οποίο προώθησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου το κίνημα των πέντε αστέρων με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους μετακινούμενους απασχολούμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτέλεσε για μας πρωταρχική προτεραιότητα και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν οι κανόνες που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στα επιδόματα ανεργίας, στα επιδόματα ασθένειας, στα επιδόματα τέκνων. Πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εδώ πέρα μια επανάσταση όσον αφορά την νοοτροπία που υπήρχε μέχρι στιγμή, και η οποία θα πρέπει σαφώς να τροποποιηθεί και να οδηγηθεί σε μία ισότιμη κατανομή των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, καθώς επίση και σε ένα σύστημα συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στα δικαιώματά τους και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αποφύγουμε καταχρήσεις και απάτες. Το να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε κοινωνικά δικαιώματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες δεν είναι κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο και διαπραγματεύσιμο με βάση την οικονομική συγκυρία που ισχύει σε μεμονωμένα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κατοχυρώνει ισότιμα τέτοια δικαιώματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες πρόσβαση στα δικαιώματα αυτά αλλά και αυστηροί κανόνε και κυρώσει όσον αφορά την παραβίαση των κανόνων αυτών. Διακόπτη πρόεδρο, Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα απλώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει τι πρωτοβουλίε αυτέ. Ολοκληρώσω, παρακαλώ πολύ, υπερβήκατε το χρόνο αγόρευση των δύο λεπτών. Η κυρία Ντεσούτερ τώρα έχει το λόγο. Äh, κυρία Επίτροπε, σας υποστηρίζουν οι πράσινοι στην εργασία που κάνετε και υποστηρίζουμε και τον ενθουσιασμό με τον οποίο επιτελέσετε την εργασία σας. Το θέμα του συντονισμού των συστημάτων ε, κοινωνικής ασφάλισης είναι σημαντικό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλούμε για Εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν με καταχρηστικές συνθήκες. Θέλουμε όλοι να είναι να απολαμβάνουν των ιδίων δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια καθήκοντα και οι ίδιες υποχρεώσεις και οι ίδιες απολαβές και κέρδη για όλους. Μιλήσατε για τον ποδηλατικό γύρο. Είπατε είμαστε λίγο πριν από το τέρμα. Είπατε ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τα επιλύσουμε. Δεν πιστεύετε όμως ότι υπάρχουν και πολιτικά εμπόδια τα οποία θα πρέπει εκτός από τα τεχνικά που μπορούμε με τεχνικού περιεχομένου λύσεις να ξεπεράσουμε, να κάνουμε κάτι για να ξεπεράσουμε και τα πολιτικά εμπόδια. Αυτά τα θέματα είναι πραγματικά μεγάλα θέματα στα οποία υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διάφορα συστήματα στις διάφορες χώρες. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, συστήματα διαφορετικά και δεν πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μία ενιαία λύση για όλους. Νομίζω ότι η Βρετανία έχει ένα σύστημα το οποίο είναι αρκετά δίκαια. Πολλοί όμως ε, πιστεύουν ότι δεν είναι σωστό και ξέρουμε ότι σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν πολλά προβλήματα και μεγάλο βάρος υφίστανται και τα σχολεία και οι γιατροί και όλοι όσοι πρέπει να παρέχονται τους επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν Κύριε Επίτροπε, ότι θα πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε, να γίνουν αλλαγές, να ε, υπάρχει περισσότερη δικαιοσύνη. Μιλήσατε για συντονισμό. Εμένα μου φαίνεται ότι μιλάμε για εναρμόνιση και πιστεύω ότι κάθε χώρα θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει και τα σύνορά της και την ομοθεσία της, αλλά η ερώτησή μου είναι ευθύντατη. Έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων τα οποία εργάζονται στον Ηνωμένο Βασίλειο η χώρα μου και θα συνεχίσει, θα συνεχίσει. Το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δικούς μας πολίτες. Ευχαριστώ. Κυρία Ροντινέλη και μετά ο τελευταίος μιλητής, ο κύριος Νικόλαος Αλαβάνος. Κύριε Επίτροπε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα θα μπορούσα να σας διηγηθώ, αν θέλετε, μια προσωπική εμπειρία. Πριν από 30 χρόνια ήμουν από τους πρώτους νέους οι οποίοι ε, συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εράσμους. Έκτοτε, μετά τις σπουδέ μου, ήθελα πραγματικά να εργαστώ σε πολλές διαφορετικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό όχι απλώς να έχω ένα αξιοπρεπή μισθό, αλλά να μπορώ πραγματικά να έχω κοινωνική κάλυψη σε οποιοδήποτε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειτο να βρεθώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό έχει να κάνει πραγματικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία υφίστανται σε κάθε χώρα. Μετά από 30 χρόνια λοιπόν, μετά την πρώτη αυτή εμπειρία στα πλαίσια του προγράμματος Εράσμους, ακούγοντάς σας σήμερα, Πραγματικά με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά και ικανοποίηση ακούω αυτά τα οποία λέτε, ότι μπορούμε πραγματικά να καταλήξουμε σε ένα συντονισμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν, αλλά να ολοκληρώσουμε την πολύ θετική εργασία που έχει ήδη επιτευχθεί. Μας ανησυχεί όμως η στάση που έχουν υιοθετήσει ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ιδίως ε, όσον αφορά τις ε, χώρες προέλευσης και την δυνατότητα καταβολής των επιδομάτων τέκνων. Τα επιδόματα αυτά θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση ποια χώρα. Αυτό έχει προκαλέσει κάποια ανησυχία. Νομίζω ότι ιδίω στο πλαίσιο των προγραμμάτων λιτότητα που έχουν επιβληθεί σε κάποιε χώρε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια απάντηση στο ζήτημα αυτό. Ο κύριος έχει το λόγο. Συναντάμε. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η νέα κυβέρνηση με επεξίδα το έργο τη προηγούμενη και τη κατευθύνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγάγει σε κεντρικό ζήτημα το ασφαλιστικό. Ακολουθώντα το σύστημα των λεγόμενων τριών πυλώνων, προτείνει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 16% για του εργοδότε, με αποτέλεσμα τη μείωση του ασφαλιστικού κόστου για τι επιχειρήσει, αλλά μείωση και τη σύνταξη για του εργαζόμενου κάποιο με 20 χρόνια ασφάλιση, για παράδειγμα, θα πάρει σύνταξη γύρω στα 380 ευρώ. Δεύτερον, ενίσχυση τη κεφαλαιοποιητική λειτουργία για την επικουρική ασφάλιση, μετατρέποντα τι φορέ των εργαζομένων σε κεφάλαιο για επενδύσει. Τρίτον, ιδιωτική ασφάλιση για συμπλήρωμα παροχών σύνταξη, μια κούρσα δηλαδή εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αλλαγέ που γίνονται στη γραμμή του Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντο, που έχει στόχο όχι την ενίσχυση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών, αλλά την απελευθέρωση χρηματοδοτικών πόρων, όπω λέει η Επιτροπή, προ τι επιχειρήσει τη Ευρώπη. Είναι γεγονό ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ο ΩΣΑ τοποθετούνται με επιφύλαξη για τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώ είναι ευπαθή σε χρηματοπιστωτικέ κρίσει και περιόδου ύβεση και έχουν οδηγήσει σε σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωση για του μελλοντικού συνταξιούχου. Ο στόχο είναι η απαλλαγή των επιχειρήσεων από το βάρο τη κοινωνική ασφάλιση. Η λογική είναι η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα υψηλότερε εισφορέ με αμφίβολε απολαυέ και πάντοτε χαμηλότερα από ό,τι πριν στη λογική τη ενεργού γύρανση και τη λεγόμενη ασημένια οικονομία. Πώ τοποθετείται η κυρία Επίτροπο για αυτά τα ζητήματα. Before I give the floor to Madam Commissioner, I just want to remind you, especially coordinators, please stay till the very end because there is... Θα του ξαναδώσω το λόγο στην ε, Επίτροπο καλώ τους συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα γιατί θα πρέπει να συνδράσουν εκ νέου συντονιστές και θα πρέπει να λάβουμε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Κύριε Επίτροπε, εσείς τώρα καλείστε να δώσετε απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα ήταν λίγο αφελές να σας ζητήσω να είστε σύντομοι γιατί μάλλον είναι αδύνατο, αλλά αν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να είστε ευσύνοπτοι στην παρεμβίασή σα. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω όντω να είμαι ευσύνοπτη και να απαντήσω ουσιοδό στα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν από του συναδέλφου. Σαφώ θα πρέπει να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αυτόν εκ των Ουκάνευ. Αλλά ξέρετε ότι έχει να κάνει και με την πολιτική βούληση. Και κατά αυτόν τον τρόπο απαντώ σε διάφορε ερωτήσει που για διάφορε ανησυχίε από διάφορου ευρωβουλευτέ και παντό και στην κυρία Ντεσούτερ. Πρόκειται για θέμα πολιτική βούληση. Σαφώ πρόκειται για ζήτημα πολιτική βούληση. Ξέρετε ότι στα πλαίσια τη πολιτική υπάρχουν ορισμένοι πολιτικοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνικά εμπόδια για να αποφύγουν να λάβουν μια καθαρά πολιτική απόφαση. Αυτή τη στιγμή όμω πρέπει να λύσουμε πραγματικά τεχνικά ζητήματα. Πώ μπορούμε δηλαδή να συντονίσουμε αποτελεσματικά τα συστήματα κοινωνική ασφάλιση έτσι ώστε όταν κάποιο μετακινείται και εργαστεί σε μία άλλη χώρα να μπορεί απρόσκοπτα να έχει πρόσβαση στα δικαιώματά του, όπως ακριβώς θα συνέβαινε και στην δική του την οικία χώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να μπορεί να γίνεται απρόσκοπτα στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος νομικής ασφάλειας και χωρίς οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιφορτίζονται πέραν του δέοντος. Πρέπει να έχουμε βέβαια τον ευκαιρό συντονισμό και τον κατάλληλο έλεγχο του συντονισμού αυτού. Ο κύριο Σμιτ βλέπω ότι έχει ήδη αποχωρήσει από την αίθουσα. Σε κάθε περίπτωση, απαντώντα του, ήθελα να του πω ότι καθότι υπήρξε υπουργό και είχε συμμετάσχει και ο ίδιο διαπραγματεύσει που έλαβαν χώρα στο Συμβούλιο, θα πρέπει εκ νέου να αναφερθούμε στο ζήτημα των μεθοριακών εργαζομένων. Και υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία ακόμα μπορούμε να διευθετήσουμε με ένα καλύτερο τρόπο σε σχέση με αυτό το οποίο προβλέπεται στην προσωρινή συμφωνία. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο βελτίωσης για το ζήτημα των μεθοριακών εργαζομένων και επ' αυτού συμφωνώ απόλυτα μετά όσα είπε ο κύριος Σμιτ. Θα προσπαθήσω να συντομεύσω κύριε Πρόεδρε. Με ρωτήσατε αν θα πρέπει να ρυθμίσουμε τον τρόπο απασχόληση των μεθοριακών εργαζομένων. Σαφώ πρέπει να το κάνουμε αυτό και κατά αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε εν γέννη τι παραμεθόριες περιοχέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί όπου υπάρχει δηλαδή η πιο έντονη κινητικότητα εργαζομένων. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να αποκομίσουμε πολύ σημαντικά διδάγματα από τι περιφέρειε αυτέ που ήδη έχουν την σημαντική αυτή εμπειρία και βέβαια Α μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διασυνοριακέ μετακινήσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητα μεθοριακέ. έτσι δεν είναι. Θα απαντήσω Ολλανδικά στον συναδελφό σας που μου έφεσε την ερώτηση Ολλανδικά ή στα Φλαμανδικά. Όπως είπε και ο κύριος Μπέγκλερ, θα πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας για το θέμα αυτό να καταβάλουμε προσπάθειες. Ξέρετε ότι ο συντονισμός των ε, συστημάτων κοινωνικής, ε, ε, κοινωνικών παροχών κοινωνικής ασφάλισης είναι δύσκολα, διότι υπάρχουν ευαίσθητα πολιτικά και άλλα στοιχεία. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως τις ε, συζητήσεις. Υπάρχουν προτάσεις λύσεων για τα περισσότερα προβλήματα. Πολλά προβλήματα έχουν ξεπεραστεί. Υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή, ας χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που μας μένει εποφελώς ώστε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Πιστεύω ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, βούληση θα μπορέσουμε πριν και να αναλάβει το έργο της η νέα Επιτροπή. Είμαι πεπισμένη διότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. Εάν υπάρχει, παραλαμβάνω, πολιτική βούληση μπορούμε να προχωρήσουμε. Μην κρυβόμαστε πίσω από την ε, ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων. Η πολιτική βούληση είναι αυτή που θα μας βοηθήσει. Τώρα, οι διάφορες ε, επιχειρήσεις λένε ότι είναι αδιαφανείς οι κανόνες, υπάρχει επαχθές αντιοικητικό, γραφειοκρατικό πλαίσιο οι εργαζόμενοι επίση ότι δεν είναι σαφή τα κριτήρια, οι εθνικές αρχές, οι υπεύθυνοι των κρατών μελών επίσης πρέπει να βοηθηθούν εάν θέλουμε να συνεργάζονται σωστά. μονο έτσι είμαι πεπισμένη ότι η, η υπεύθυνη Ευρωπαϊκή Αρχή σε θέματα εργασιακά θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και να βοηθήσει πολύ. Και θα πρέπει να θα αρχίσουμε ήδη το, με κάποιες δραστηριότητες τον Οκτώβριο και είμαι σίγουρη ότι έτσι θα υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών. Υπάρχουν όμως και προβλήματα χρόνου προσθεσμιών που πρέπει να σεβαστούμε. Μου είπατε πού υπάρχουν οι διαφωνίες, ποιες χώρες είναι αυτές που δεν μπορούν στο Συμβούλιο να υπερψηφίσουν. Υπάρχουν κράτη-μέλη που υπερψήφισαν, αλλά είχαν προβλήματα, διότι καμία λύση δεν είναι 100% τέλεια, σύμφωνα με τις επιδημίες του καθενός. Έτσι όμως είναι η Ευρώπη. Είμαστε 28, ίσως το μέλλον 27, δεν ξέρουμε, αλλά πάντα πρέπει παρά τις διαφωνίες να συμφωνούμε. Το ίδιο κάνετε και εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο, το ίδιο, κάνουν, το ίδιο κάνουν, γίνεται και σε επίπεδο Συμβουλίου και εμείς στην Επιτροπή ακούγοντας όλους από τα κράτη-μέλη, τους εκπροσώπους, προσπαθώντας να καταλάβουμε και να καταθέσουμε προτάσεις που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και στην εμπειρία του καθενός. Δεν μπορώ λοιπόν να σας πω ρητά που βρίσκονται οι διαφωνίες, αλλά πρέπει να πω ότι οι περισσότερες χώρες θέλουν πραγματικά να καταλήξουμε σε συμφωνία και να βρούμε λύσεις, διότι είναι απαραίτητο. Το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έκαναν ε, θετικές προτάσεις και αποτίμηση του τι κάναμε μέχρι τώρα και να συνεχίσουμε. Τώρα, στη, στα πλαίσια της προειδοποίησης, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάντα για τις διάφορες επιχειρήσεις ε, ε, κάτι το οποίο πρέπει να δίδεται απαραίτητα στα διάφορα επαγγελματικά ταξίδια, στις διάφορες μετακινήσεις για, για λόγους εργασίας για λίγες μέρες. Δεν πρέπει να έχουμε αυτή τις προειδοποιήσεις ότι, ότι κάποιος δηλαδή καλύπτεται από το σύστημά του αν φύγει κάποιες μέρες από την άλλη. Με πάρα πολύ εύκολο τρόπο τώρα μπορούμε να το λύσουμε αυτό το, το πρόβλημα και μπορούμε να σας δώσουμε τους σχετικούς ορισμούς γιατί χρειάζομαι πάρα πολύ χρόνο τώρα να σας το εξηγήσω θα πρέπει να κοιτάξω και όταν γραφάμε αλλά πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχουν μεγάλες βελτιώσεις Βεβαίως δεν μπόρεσαν όλα τα κράτη-μέλη να το συζητήσουν αυτό το θέμα διεξοδικά, αλλά θα φαντάζομαι ότι θα βρούμε μια καλή λύση η οποία θα αρμόζει σε όλους. Επίσης, Επίσης ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης, όπως υπόθηκε, είναι ένας τρόπος να υποσκάψουμε τα συστήματα των κρατών μελών. Αυτό δεν ισχύει και είμαι ξεκάθαρη και ε, πολύ αυστηρή αυτό. Ο συντονισμός δεν είναι εναρμόνιση. Κάθε κράτος μέλος έχει την ελευθερία να οργανώσει το σχέδιο και τον τρόπο χρηματοδότησης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που διαθέτει. Αυτό είναι μία αρμοδιότητα των κρατών μελών, θα παραμείνει ε, εσαΐ και δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι σύμφωνα με τις, που ισχύει σύμφωνα με τις συνθήκες, η αρχή της επικουρικότητας δηλαδή. Το θέμα όμως είναι ότι όταν ε, οι εργαζόμενοι μετακινούνται, όταν ε, μετατίθενται εργαζόμενοι, όταν οι εργοδότες στέλνουν κάποιον σε κάποια άλλη χώρα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι επιπτώσεις σε επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης και πρέπει να πούμε, να συμφωνήσουμε ποιο σύστημα θα εφαρμόζεται την κάθε στιγμή. Δεν αλλάζουμε το περιεχόμενο του συστήματος, ούτε το σχέδιο ούτε τον τρόπο που θα χρηματοδοτούν τα κράτη-μέλη τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Συντονισμός ε, είναι μία λέξη που σε κάποιες γλώσσες ίσως να ακούγεται το ίδιο με την εναρμόνιση, όμως είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ωραία, τι άλλο έχουμε. Ναι, και η ερώτηση για τη μείωση των, ε, της δύναμης των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ε, όχι, δεν θέλουμε να το κάνουμε πιο φθηνό για τις αρχές. Θέλουμε μια βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ε, έρχομαι από το G20 στην Ιαπωνία. Είδα πολλά κράτη, πολλά κράτη στον κόσμο που μας μίλησαν για το ίδιο πρόβλημα, τη γύρανση του πληθυσμού. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπω περισσότερο σε αυτό το θέμα. Και νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι με αυτόν τον τρόπο έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Είναι και λίγος ο χρόνος. Ναι, φυσικά, για το Ηνωμένο Βασίλειο όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες. Αν έχουμε ένα τακτικό Brexit, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια μεταβατική περίοδο και θα ε, γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώματα, όπως και τώρα. Θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι αρχές που ισχύουν ήδη. Τα υπόλοιπα θα εξαρτηθούν από τη μελλοντική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου για αυτά τα δικαιώματα. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Τώρα, αν γίνει Brexit χωρί συμφωνία, Όλα θα βασιστούν στα μέτρα έκτακτης ανάγκης. Φυσικά θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες που έχουν δικαιώματα σε, ε, θεμελιωμένα. Ε, ελπίζω ότι για το μέλλον θα βρούμε μια καλή συμφωνία και δεν θα έχουμε ένα άτακτο Brexit. Ελπίζω ότι ε, δεν θα συμβεί και δεν είναι και το θέμα της σημερινής συνάντησης. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά αξίζεται χειροκρότημα, κύριε Επίτροπε. ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω ότι είστε όλοι ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις που σας έδωσε η Επίτροπος και πραγματικά απάντησε η Επίτροπος σε όλες τις ερωτήσεις μας. Ήρθε η ώρα τώρα για τη συνεδρίαση των συντονιστών και θα κληθούμε να πάρουμε την κατάλληλη απόφαση όσον αφορά την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Και κάτι ακόμα. Η Πρόεδρος ευχαριστεί τους διερμηνείς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή σας εργασία, λέει η Πρόεδρος. Ποιον άλλον από μένα να ευχαριστήσω. Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίας των στονιστών, όπου θα έχουμε διερμηνία στα γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και πολωνικά.